των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς Μεταφορής. Είναι το θέμα που θα εξετάσουμε τώρα. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κράμερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να κάνω μια ερώτηση στην Επιτροπή όσον αφορά το θέμα του περιορισμού λόγω των ε, ρουσικών ε, αποφάσεων και των αντίκτυπων αυτών των περιορισμών Witamy panią komisarz. Panie pośle, może pan kontynuować. Bardzo proszę. Μπορείτε να συνεχίσετε. Καλωσορίζουμε τον Επίτροπο. Θα ξαναρχίσω κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού θέτει την εξής ερώτηση για τον αντίκτυπο των περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορής. Στις 7 Αυγούστου 2014 η Ρωσική Ομοσπονδία επέβαλε απαγόρευση για την εισαγωγή ορισμένων τροφίμων και γεωργικών προϊόντων κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον τομέα των μεταφορών αυτός ο αποκλεισμός σημαίνει την απαγόρευση της εισόδου οχημάτων μεταφέρουν γεωρικά προϊόντα και τρόφιμα και αυτό βεβαίως οδηγεί σε μεγάλη απώλεια συμβάσεων. Η Ρωσική Ομοσπονδία παρακολεί την διεκπαιρέωση και τη διαμετακόμιση προς τρίτες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη ζητάει εποπτεία ε, για την ε, μεταφορά από την επικράτειά της τροφίμων και υγειογικών προϊόντων. Αυτό αυξάνει σημαντικά το κόστος. Η ρωσική αγορά είναι οικονομικά ελκυστική, ιδιαίτερα για εκείνους που είναι εγκατεστηλημένοι σε χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, συνορεύουν με τη Ρωσία. Η Επιτροπή έχει ήδη αντιδράσει στους ρωσικούς περιορισμούς θεσπίζοντας βροχυπρόθεσμα μέτρα για τη στήριξη της αγοράς που ξεπερνούν τα 155 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ε, δυσκολιών ιδιαίτερα στην αγορά που αφορούν τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο οι επιπτώσεις στην αγορά μεταφορών έχουν ε, πολύ λιγότερο ληφθεί υπόψη και κυρίως αναφερόμαστε εδώ σε βιομηχανικά προϊόντα και σε τρόφιμα που μεταφέρονται κατά κύριο λόγο οδικός. Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις μεταφορικές που εξειδικεύονται στα τρόφιμα και που πλήττονται σήμερα σημαντικά από τον ρωσικό εμπορικό αποκλεισμό, χάνοντας σημαντικές συμβάσεις. Επιπλέον βλέπουμε ότι στις 25 ε, και 26 Σεπτεμβρίου του 2014 το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών ITF που έλαβε χώρα στο Παρίσι αναφέρθηκε στα προβλήματα αυτά και της μεταφοράς εντός επικράτριας της Ρωσίας και από την 1η Ιανουαρίου του 2015 βλέπουμε ο αριθμός των αδειών Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών που ισχύουν επί του ρωσικού εδάφους έχουν περάσει από 67 σε 16. Η ερώτηση λοιπόν είναι εξής. Που το πρίσμα των η Επιτροπή είναι ενήμερη για την σοβαρότητα αυτής της κατάστασης και για το σύνολο των επιπτώσεων από αυτόν τον ρωσικό αποκλεισμό στους μεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε η Επιτροπή να μας παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις απώλειες αυτές στον τομέα των μεταφορών. Τρίτον, Ποια είναι τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, προτίθεται να λάβει η Επιτροπή έτσι ώστε να εξισορροπηθεί αυτή η απώλεια που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, πώς προτίθεται η νέα κυβέρνηση να παρέμβει στον τομέα των μεταφορών και των επιπτώσεων αυτών, ιδιαίτερα για αυτούς που πλήττονται από αυτών των αποκλεισμών. Και πέμπτον, προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει δράση στα πλαίσια της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής, προκειμένου να καταθέσει καταγγελία εναντίον της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Κράμερ εκ μέρους της Επιτροπής. επίτροπο Επίτροπος, μπορείτε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη, η ρωσική απαγόρευση της εισαγωγής ορισμένων αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κάποιες άλλες χώρες είχε αντίκτυπο στο κλάδο των αγροτικών αλλά και τις οδικές μου μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σε χώρες που έχουν πολλές ε, γεωργικές εξαγωγές προς τη Ρωσία. Πριν την θέση σε ισχύ της ρωσικής απαγόρευσης, η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά της ΗΠΑ. Από πλευράς αξίες, οι μισές ε, εξαγωγές ύψους 5,1 δις ευρώ πλήττονται από τη ρωσική απαγόρευση. Όλα αυτά κυρίως αφορούν στα κρέατα, τα προϊόντα κρέατος, το γάλα, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια, τα θαλασσινά και τα νοπά οποροκυπευτικά. Και επίσης πλήττεται και η διαμετακόμιση αυτών των προϊόντων με κατεύθυνση την Ασία από τη στιγμή που πρέπει να περάσουν από τη Ρωσία. Και άρα επεκτείνεται η απαγόρευση και στις ευρωπαϊκές εξαγωγές ε, τέτοιου είδους προϊόντων προς τις χώρες της Ασίας. Οι οδικές μεταφορές είναι και η βασική ε, δίωδος, ο βασικός διάβλος μεταφορών. Το των γεωργικών εξαγωγών από Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία μεταφέρεται ε, οδικός και από πλευράς όγκου και από πλευράς ε, τιμών και ποσοτήτων. Επομένως, Πέρα από την ε, παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι οδικοί μεταφορείς πλήττονται ιδιαιτέρως από τη ρωσική απαγόρευση. Και εγώ και η ομάδα μου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό, το συνειδητοποιούμε πλήρως. Ε, πόσο υποφέρουν. Είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Εξαρτάται από τις ε, κατατόπους περιστάσεις και συνθήκες. Πολλά από τα απαγορευμένα αγαθά τα οποία θα είχαν εξαχθεί στη Ρωσία τώρα επανακατευθύνονται και πολλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις η τιμή των προϊόντων έχει, έχει πέσει δραματικά λόγω της υπερπροσφοράς που έχει δημιουργηθεί με την απαγόρευση αυτή. Και μάλιστα οι οδικοί μεταφορεί που ειδικεύονται στι εξαγωγέ γεωργικών προϊόντων στη Ρωσία και που έχουν κάνει μεγάλε επενδύσει σε εξοπλισμό όπω είναι τα οχήματα, τα φορτηγά με ψυγεία θα αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν ενδεχομένω πάρα πολλέ δυσκολίε. Αυτό βεβαίω εξαρτάται από το πόσο καλά κατάφεραν να επανακατευθύνουν το στόλο τους αλλού. Και βεβαίως οι μεγάλες ε, ενταλίκες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από όλους τα πολύ μεγάλα φορτηγά. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Αντίθετα με τους συναδέλφους μου που ασχολούνται με το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας, εγώ δεν έχω ταμείο επίγουσας βοήθης ή προήθειας ε, που να δώσω στους εθνικούς μεταφορείς. Μπορούν ε, να τύχουν λοιπόν ενδεχομένως κρατικών ενισχύσεων. Οι ελάχιστοι κανόνες επιτρέπουν κρατικές ενισχύσεις 100.000 ευρώ σε βάθος χρόνου τριών ετών. Υπάρχουν κάποιοι όροι και προποθέσει που πρέπει βεβαίω να τηρούνται, αλλά μέχρι 100.000 ευρώ για τρία χρόνια δεν χρειάζεται να κοινοποιηθεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί το κράτο να τα δώσει. Και η κρατική ενίσχυση είναι μια επιλογή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό ε, πολύ αυστηρέ ε, ε, προποθέσει και άνω των 100.000 ευρώ θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι οδικέ μεταφορέ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και και Ρωσίας διέπονται από διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας και του εκάστοτε κράτους μέλους. Άρα τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία πρέπει να εξετάσουν αυτό το θέμα και να δουν τι καλύτερο μπορούν να κάνουν επί τη βάση των διμερών συμφωνιών. Δεν έχουμε ε, σχετική συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε έχουμε ανοίξει τέτοιου είδους διάλογο. Αυτό βέβαια μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσουμε και να το χειριστούμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά το κατά πόσο είναι συμβατοί οι περιορισμοί που επιβάλλει η Ρωσία με τον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού και της απαγόρευσης ε, της εισαγωγής και της διέλευσης αυτών των προϊόντων στη Ρωσία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για αυτή την τόσο σημαντική παρέμβαση. Ξεκινάμε τις πολιτικές ομάδες για το ΕΛΚΕ. Η κυρία Λούκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η Ρωσία απαγορεύει τις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγώντα σε επιδείνωση τις κατάστασεις σε πολλές επιχειρήσεις ε, γεωργικές, μεταποίησης αλλά και στις μεταφορές. Η απαγορεύση των μεταφορών οδηγεί σε αδυναμία διέλευσης των οχημάτων ε, από τη ρωσική επικράτεια με μεγάλες ζημίες και κίνδυνο πτώχευσης ορισμένων μεταφορικών εταιριών. Πέραν της οικονομικής πτυχής δεν πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνική ανεργία για πολλούς ανθρώπους που αργά γρήγορα θα χρειαστούν επιχορηγήσεις κάποια οικονομική ή κοινωνική υποστήριξη. Πολλοί παραγωγής εμπορευμάτων που εξάγονται στη Ρωσία, πολλοί ιδιοκτήτε μεταφορικών εταιριών και εξαρτώμενοι από αυτούς βρίσκονται υπό αυτή την απειλή. Αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τις πολωνικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Είναι σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρούμε λύσεις που θα οδηγήσουν στην επαρκή υπεράσπιση των πληγέντων. Η έλλειψη μηχανισμών αντιμετώπισης αυτού του εμπάργου θα μπορούσε να οδηγεί σε δυσκολίες ε, στην αγορά των ευρωπαϊκών μεταφορών. Η Πολωνία είχε προτείνει λύσεις συγκεκριμένες στο Συμβούλιο για υποστήριξη προς μεταφορικές εταιρείες που είναι θύματα του ρωσικού εμπάργου. Όπως για παράδειγμα διαφορετικό δίκτυ για τη δυνατότητα δημόσια στήριξης ή στήριξη και ορισμένες επιχειρήσεις ε, ε, ε, σε εθελοντική βάση το γνωρίζει, τα γνωρίζει αυτά τα προβλήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν τα γνωρίζει τι συγκεκριμένες λύσεις προτείνει, ποια βοήθεια η βοήθεια που αναμένεται από όλους αυτούς που φοβούνται την ανεργία και την απώλεια και, τη, και τις ζημίες που μπορεί να υποστούν. Εκ μέρους των σοσιαλιστών ε, τα παρδέλια λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σε μια παγκόσμια οικονομία τα εμπορεύματα διακινούνται διαρκώς μέσα σε πολύ περίπλοκα δίκτυα σε σε γεωγραφικές περιοχές. Η απαγόρευση των γεωργικών προϊόντων από τη Ρωσία, προϊόντων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας ε, δείχνει πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει μια τέτοια πολιτική απόφαση σε διάφορους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταθώ στο πλάι όσων εφιστούν την προσοχή στις συνέπειες που έχουν όλα αυτά για τη τομέα των μεταφορών. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης αν δεν αντιληφθούμε τις σοβαρές οικονομικές ζημιές λόγω συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και χαθεί ε, από τις μεταφορικές εταιρείες. Είναι πολλά τα γεωργικά προϊόντα, είναι μεγάλο το κόστος για τους γεωργούς και για τους μεταφορές. Ε, επηρεάζεται ολόκληρη η οικονομία, όχι μόνο ένας ή άλλος τομέας. Λόγω της εσωτερικής αγοράς, οι επιπτώσει γίνονται στη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να μα παράσχει επαρκή δεδομένα όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτή τη απαγόρευση, ώστε μαζί να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το ECR ο κύριος Πόρεμπα αντιπρόεδρος μας της Επιτροπής Μεταφορών Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, bardzo e, dziękuję za możliwość w tej ważnej sprawie, bo myślę, że... Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που συζητούμε σήμερα και νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι ότι η απαγόρευση, ο αποκλεισμό από τη μέση τη Ρωσία πλήττει και τα γεωργικά προϊόντα αλλά και τον τομέα των μεταφορών. Πρόκειται για μία στρέβλωση, καθότι δεν πλήττεται μόνο μία χώρα. Δεν πρόκειται για ένα τοπικό θέμα, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Λετωνία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ελλάδα και η χώρα μου, η Πολωνία, έχουν σημαντικές απώλειες από τον Αύγουστο του 2014 όταν ξεκίνησε αυτή η απαγόρευση οι απώλειες στον ε, τομέα των μεταφορών της Πολωνίας ξεπερνούν τα 22 εκατομμύρια ευρώ και 48 τον Νοέμβριο. Έφτασε αυτό το ποσό. Η Ρωσική Ομοσπονδία εμποδίζει την μεταφορά προϊόντων, εμπορευμάτων μέσα από την χώρα. Δεν υπάρχει όμως κανένας τρόπος να αντιτεθούμε σε αυτό. Ελέγχουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μεταφορικές επιχειρήσεις, τους απαγορεύουν το πέρασμα και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα αντίστοιχο προς τις ρωσικές επιχειρήσεις. Δεν αντιδρούμε λοιπόν με αντίστοιχα αυστηρό τρόπο και βρισκόμαστε αποκλεισμένοι και σε αντιέξοδο. Σήμερα βλέπουμε παραδείγματος χάρη στην Γερμανία να υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια για το πέρασμα των δικών μας ε, μεταφορών κάτι που επίσης πλήττει πολύ τις επιχειρήσεις μας και από την άλλη πλευρά έχουμε την απαγόρευση τον αποκλεισμό από μέρος της Ρωσίας. Σας παρακαλώ πολύ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πλήττονται πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάιστερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δώσατε την απάντηση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να κάνετε κάτι εσείς. Εμείς ε, βεβαίως δεν ε, θέλουμε εδώ να εκφραστούμε για τις κυρώσεις. Την Τετάρτη θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε με ποιον τρόπο με την επιβολή των κυρώσεων. Το θέμα είναι όμως να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα αυτών που έχουν πληγεί. Έχουμε συζητήσει για τον αγροτικό τομέα, για την δυνατότητα να στηρίξουμε τον τομέα αυτό, αλλά τίποτα δεν έχουμε πει για τον τομέα των μεταφορών. Ξέρουμε ότι όλα αυτά τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα μεταφέρονται μέσα σε ψυγεία, σε οχήματα. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές να βρουν άλλες αγορές για να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Οι άλλες αγορές όμως θα πρέπει να δούμε ποιες είναι και θα πρέπει να δούμε εάν τελικά αυτές οι χώρες εποφελούνται από αυτήν την απαγόρευση της ε, Ρωσίας, ε, τον αποκλεισμό της Ρωσίας και θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση και βεβαίως επειδή πολλά μέσα δεν έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και οι ίδιες οι χώρες να δουν τι μπορούν να κάνουν. Σήμερα μιλάμε για μια ενιαία αγορά, για μια εσωτερική αγορά η οποία θα πρέπει να αντιδράσει με αλληλεγγύη προς αυτούς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο. Μιλήσαμε για τις κυρώσεις αλλά σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση, μια λύση η οποία να εξισορροπεί την κατάσταση και η οποία να βοηθάει τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν πληγεί να ανασάνουν. Γιατί αλλιώς θα αυξηθεί το συνέστημα της αδικίας. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση που να είναι δίκαιη και για τον τομέα των μεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου προς την Κομισιόν, την οποία συζητούμε σήμερα, δείχνει ότι στην αίθουσα αυτή υπάρχει επιλεκτική μνήμη. Η Επιτροπή μας κάνει λόγο για τα μέτρα περιορισμού εισαγωγών και μεταφορών αγροτικών προϊόντων που έλαβε η Ρωσία στις 7 Αυγούστου 2014, ξεχνώντας ότι αυτά αποτελούσαν απάντηση στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της ρωσίας σχετικά με την ουκρανική κρίση λίγες μέρες νωρίτερα στις 31 Ιουλίου. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι οι συνάδελφοι της Επιτροπής Μεταφορών επικαλούνται τώρα και τις απαγορεύσεις επιβολής περιορισμών στη διακίνηση αγαθών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αν όμως κάποιος έχει παραβιάσει πρώτος τις ρυθμίσεις του οργανισμού, αυτός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ο κανονισμός 833 του 2014 περί κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ούτε καν μνημονεύει συγκεκριμένα και μάλιστα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης ή των μελών της που θίγονται από ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανική κρίση ώστε να δικαιολογείται η επιβολή των κυρώσεων. Η ουσία είναι ότι οι κυρώσεις έχουν αποδειχθεί ατελέσφορες για να επηρεάσουν τη ρωσική πολιτική και το μόνο αποτέλεσμα του εμπορικού πολέμου είναι να ζημιώνονται ευρωπαίοι παραγωγοί και μεταφορείς. άρα ή θα πρέπει να αρθούν αμοιβαία τα μέτρα ή αλλιώς η ευρωπαϊκή ένωση να καταβάλει πλήρεις αποζημιώσεις στους θυγόμενους για όσο χρόνο εξακολουθεί να καταβαλει πληρεις αποζημιωσεις στους στιγομενους για οσο χρονο εξακολουθει να ισχυει ο κανονισμός 833 του 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούνκριν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, είναι σαφές, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Είναι ένα πρόβλημα που πλήττει πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν τρόφιμα ή γεωργικά προϊόντα. Και ξέρουμε από πού προέρχεται. Ξέρουμε από τι εξαρτάται είναι το προϊόν έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κανείς να υπολογίσει και να εκτιμήσει τους λόγους αρκετά εύκολα. Και είναι επίσης σαφές ότι τα κράτη-μέλη που έχουν ισχυρό κλάδο μεταφορών προς τη Ρωσία πλήττονται περισσότερο από άλλα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αλλάξει αυτό. Το έχει επιβεβαιώσει και η Επίτροπος Τροποντινά. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι τελικά ότι το γεγονός ότι οι μεταφορείς που πλήττονται περισσότερο είναι αυτοί που επένδυσαν σε φορτηγά ψυγεία. Έκλεισε η ρωσική αγορά και έχουν πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μου. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύσει αυτό το πρόβλημα. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, έχουν, να έχουμε μεταφορείς που έχουν επενδύσει στα μέγα φορτηγά Σουηδούς μεταφορείς που επένδυσαν σε αυτά τα φορτηγά για να μειώσουν το κόστος και να είναι ανταγωνιστικοί και δεν μπορούν τελικά να δουλέψουν και να λειτουργήσουν. Δεν δουλεύει η εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μαρή Κριστίν Ανατού, μια εγγεγραμμένη για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πάω να εκπλήσουμε το έμπαρκο της Ρωσίας για τα τρόφιμα από Ευρώπη επιβλήθηκε στις 6 Αυγούστου 2014 ενώ οι πρώτες κυρώσεις είναι τις 17 Μαρτίου του 2014. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν από τις Βρυξέλλες 6 φορές μέχρι την 31 Ιουλίου του 2014. Το Front National αντιτέθηκε από το Μάρτιο σε αυτές τις κυρώσεις, κρίνοντας τις ακατάλληλες, αναποτελεσματικές και επικίνδυνες για τις οικονομίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό δείχνει καθαρά ότι το Front National είχε ε, Δίκιο που αντιτέθηκε το ρωσικό εμπάργο ήταν ε, μια σωστή δίκαιη απάντηση της κυρίως Ευρωπαϊκή Ένωσης. Οι οδικές μεταφορές λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα πρώτα θύματα των παράλογων κυρώσεων των Βρυξελών. Αντί λοιπόν να διαμαρτύρομαι για τις ε, επιπτώσεις τους όπως έκανε ο κύριος Κράμερ θα προτιμούσα να ζητήσω από την Κομισιόν να άρει αυτές τις κυρώσεις και ε, με αυτόν τον τρόπο θα αρκεί το δικό του το εμπάργο. Ε, do accept a Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κράμερ. Κύριε Κράμερ, παρακαλώ. Micro, Nur darauf hinweisen, ist Ihnen das als... Να πω ότι είστε σαν πρόεδρος της Επιτροπής και δεν ήταν η άποψη η δική μου η προσωπική, αλλά άσχετα με αυτό θέλω να σας πω ότι αν ξεκινήσετε αυτή την ιστορία, ξεκινήστε με το ότι η Ρωσία καταρχήν έκανε την πρώτη παραβίαση με αυτά που έγιναν στην Κρυμαία και ξεκινήστε την ιστορία από την αρχή και κατόπιν ακολούθησαν οι κυρώσεις. Κύριε Κράμερ, κατάλαβα πολύ καλά με ποια ιδιότητα μιλήσατε και γνωστή είναι η ιστορία. Ξέρω πολύ καλά ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν εδώ και όταν κάποιος παρεμβαίνει στην εθνική κυριαρχία κάποιων άλλων κρατών συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και αυτό έγινε και με τη Ρωσία εξάλλου. Ο κύριος από το ΕΛΚΙΑ δύο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρεμβαίνω μετά από τη συνάδελφο του Front National ε, γιατί μπορούμε να δούμε έτσι καθαρά τις διαφορές. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει λόγω μιας διένεξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Στην Ευρώπη επιλέξαμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη διένεξη με κυρώσεις οι οποίες πλήττουν πολλούς οικονομικούς ε, τομείς ε, στην Ευρώπη που αισθάνονται τις αρνητικές επιπτώσεις των κυρώσεων αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το όσο είπε ο συνάδελφος ο κ. Κράμερ οι διεθνεί ε, συνθήκες πρέπει να γίνονται σεβαστές. Εννοείται δεν είναι εύκολο η Επίτροπος έχει δίκιο η Γεωργία έχει δικούς τους δικά της κονδυλία παρέμβασης που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε τον τομέα των μεταφορών στην Πολωνία για παράδειγμα οι Πολωνοί συναδέλφοι υποφέρουν λόγω αυτών των κυρώσεων είναι κρίμα που η Επιτρόπος δεν κάνει κάτι παραπάνω παρα, παραθέτει μόνο τα γεγονότα δεν μας προσφέρει καμία λύση να σας κάνω τρεις ερωτήσεις λοιπόν τι επαφές έχετε εσείς με την κυρία Μογκερίνη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά ε, κονδύλια για επίγοντα περιστατικά. Δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον τομέα των μεταφορών στην Πολωνία. Έχουμε το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση που έχει πολλά χρήματα. Χρησιμοποιείται για τις βιομηχανικές αναδιαρθρώσεις. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τον τομέα των μεταφορών. Και μετά το σημαντικό ερώτημα του συνάδελφου του κ. Κράμερ. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Θα υπάρξει κάποια επίσημη διαμαρτυρία ε, για τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κύρκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η δίκαιη επιβολή του εμπάργου στη Ρωσία λόγω των γεγονότων στην Κρυμαία και την υπόλοιπη Ουκρανία και η απάντηση της Ρωσίας δημιούργησε τα γνωστά μεγάλα προβλήματα στο εμπόριο κυρίως αγροτικών προϊόντων τόσο στην ελλάδα όσο και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. αυτό που είναι λιγότερο γνωστό στους πολίτες είναι το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον κλάδο των μεταφορών μόνο για την ελλάδα υπολογίζουμε δέκα εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση διαφυγόντα κέρδη. καταλαβαίνετε πως μέσα στην τεράστια κοινωνική κρίση που περνάει η ελλάδα και σε συνθήκες πολλές φορές αθέμητου ανταγωνισμού η κατάσταση αυτή μπορεί να αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα η απάντηση της επιτροπής ότι το δεκέμβριο του 2014 που αρνείται κάθε βοήθεια και προτρέπει τον κλάδο να προσαρμοστεί σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο ακούγεται ως κοροϊδία. φυσικά αυτό κάνουν οι άνθρωποι αλλά η απόλυση εισοδήματο λόγω μιας πολιτικής απόφασης ολόκληρης της ένωσης πρέπει με κάποιο τρόπο να αντισταθμιστούν αλλιώς πρόχουμε τους πολίτες να προσλαμβάνουν αρνητικά τις πολιτικές μας. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζήλε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν θέλουμε εμείς εδώ να παραπονεθούμε γενικώς επειδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα από μέρους της Ρωσίας. Έτσι και αλλιώς οι κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν γιατί ξέρουμε ότι η αντίδραση της Ρωσίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση εμείς να υποχωρήσουμε από τη στιγμή που πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Βεβαίως πλήττονται σήμερα οι μεταφορείς μας και βλέπουμε ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αυτές τις πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις. Πρέπει να στηρίξουμε τους μεταφορείς μας και οι περισσότεροι μεταφορείς από την Ανατολική Ευρώπη πλήττονται σήμερα κυρίως από το dumping Ξέρουμε παραδείγματος χάρη και τι επέβαλε η Γερμανία που επίσης είναι ένα επιπλέον βάρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ σοβαρά είναι κυρίως στη Λιθουανία διότι το 5% του ε, πληθυσμού που εργάζεται απασχολείται σε αυτό το κλάδο. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για εμάς και χρειαζόμαστε τη συνεισφορά σας, τις ιδέες σας, πώς θα επιβιώσουμε γιατί εμάς χτύπησε ε, αυτός ο τυφώνας τελικά. Ε, προστρέχουμε σε εσάς για βοήθεια. Θέλουμε να είστε δημιουργικοί, να βρούμε τη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Και κοιτάξτε και τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Γερμανία τελικά ψήφισε βασικό μισθό και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε εμείς, γιατί δεν είμαστε τόσο πλούσιοι όσο οι Γερμανοί. Το ίδιο και η Γαλλία και το Βέλγιο. Θέλουν οι οδηγοί να κοιμούνται σε ξενοδοχεία που δεν υπάρχουν. Ας ενωθούμε για να αλληλοβοηθηθούμε, να μην ε, κατασπαράζει ο ένας τις άρκες του άλλου. Ας τα ενωθούμε για να αντιταχθούμε μαζί στη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Τσιλσίμα. Θα ήθελα να τονίσω τον αντίκτυπο στο εμπόριο που έχει το θέμα των απαγορεύσεων της Ρωσίας. Ε, ξέρετε, οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να κάνουν σωστές επιχειρηματικές, δεν μπορούν να έχουν σωστές επιχειρηματικές σχέσεις με τη Ρωσία και τώρα πρέπει να τύχουν στηρίξεις από τους φορολογουμένους. Έχουμε αγρότες που δεν έχουν αγορές να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Πριν από το εμπάργκο, το 5% των εξαγωγών ε, γινόταν οδηγός. Ο αντίκτυπος σε όλους αυτούς τους κλάδους της οικονομίας δεν πρέπει να υποτιμηθεί γιατί είναι τεράστιο το έξτρα κόστος και αυτό αυξάνει τη τιμή των προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για αυτές τις αστάθειες. Ήταν λάθος η επέκταση προς Ανατολάς, η πολιτική και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυπάται βαθιά για τις πράξεις του. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχετε μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Από τον κύριο Γιάκοφτσιτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξής. Μιλήσατε πολύ άσχημα για τις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τις χώρες που πρόσφατα έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλήσατε πολύ άσχημα και για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν τρέπεστε να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για αυτές τις χώρες και για αυτούς τους λαούς που ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ήλπιζαν ότι θα ζήσουν σε μια ενωμένη Ευρώπη. Θέλετε να απαντήσετε λέει ο Πρόεδρος ή όχι. Καλώς. Ο κύριος Σαλίνη παρακαλώ, από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Επιτρόπε. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ σήμερα τόσο αργά το βράδυ για να συζητήσουμε σημαντικά ζητήματα στη δική μου χώρα. Οι επιπτώσεις από αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν λιγότερες διότι η Ιταλία ε, αντίθετα από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, που δικαίως ε, αναφέρονται σε αυτό το πρόβλημα έχει διαφορετικές συνθήκες αλλά θα συμμετάσχουμε συμμερίζομαι με τα προβλήματα όπως παρουσιάστηκαν από τον κύριο Κράμερ και συμμερίζομαι τις ανησυχίες και των υπολείπων συναδέλφων με κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποφύγει την υποχρέωση της να δώσει κάποια απάντηση και για το ζήτημα των οδικών μεταφορών που όπως υπενθυμίσατε ότι ένα μέσο όπου δεν προβλέπονται συγκεκριμένε παρεμβάσει υποστηρικτικέ ε, ε, για τι ζημίε που έχουν υποστεί οι επιχειρηματίε σε αυτόν τον τομέα. Και αύριο θα ξαναμιλήσουμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα για το ενδεχομένου οικονομικής ε, αρρωγής ε, σε περίπτωση σημαντικών οικονομικών προβλημάτων σε επιχειρήσεις στην Ευρώπη όπως στον τομέα της ε, όπως και στην Γεωργία που αναφέρατε εσείς δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τον τομέα των μεταφορών όπως είπε κάποιος θα πρέπει να επινοήσουμε κάποια απάντηση, κάποια απόκριση ε, από τέτοιες μικρές αποκρίσεις φάνταστες μπορεί να αναγεννηθεί η ελπίδα η μόνη δυνατότητα που έχουμε να αποφεύγουμε συζητήσεις παράξενες όπως ακούσαμε πριν από λίγο με στις οποίες ψάχνουμε να βρούμε ποιος στέει ποιο ε, επέβαλε πρώτα τι κυρώσει και ποιος, αν ο άλλο επέβαλε πρώτα το εμπάργκο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να βρούμε απαντήσει για ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη που υπάρχει σήμερα. Το πρόβλημα των οδικών μεταφορών είναι συγκεκριμένο Αυτό πρόβλημα στο οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε να παρέμβουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Ντεμόντε. Ιζαμπέλα Ντεμόντε για ένα λεπτό, παρακαλώ. Η Ρωσική Ομοσπονδία απαγόρευσε την οδική εισαγωγή κάποιων εμπορευμάτων και αυτό δημιουργεί ζημιά σε πολλούς τομείς. Όχι μόνο στους γεωργούς που υποχρεούνται να αφήνουν ε, τόνους εμπορευμάτων αλλά και τις ε, εταιρείε οδικών μεταφορών που μετέφεραν τα προϊόντα αυτά για τις οποίες ακυρώθηκαν σημαντικές ε, συμβάσεις. Παρότι υπάρχουν, έχουν προβλεφθεί οικονομικές βοήθειες για τον τομέα της γεωργίας, για τις οδικές μεταφορές, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ενώ αυτή πλήττεται εδώ και χρόνια από την κρίση που πλήττει την Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση για να βοηθήσουμε ένα τόσο σημαντικό τομέα για την οικονομία μα με συγκεκριμένε παρεμβάσει για να καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικέ τι οδικέ μεταφορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σλοτόφσκι από το ECR έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, σύμφωνο με όλους όσους μίλησαν για το θέμα αυτό, αναφερόμενοι στις κυρώσεις της Ρωσίας, που είναι το αποτέλεσμα των δικών μας κυρώσεων. Από τις δικές μας όμως κυρώσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από ένα έγκλημα. Η φίλοι από το Εθνικό Μέτωπο μίλησε για το θέμα αυτό λέγοντας ότι το θέμα μπορεί να λυθεί πολύ απλά. Κοιτάξτε, πριν από 200 χρόνια ξεκίνησε μία τέτοια παρόμοια επίθεση της Ρωσίας στην χώρα μου. Αλλά ήθελα να σας πω ότι αυτές οι επιθέσεις έχουν επιπτώσεις και κόστος και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτή την κατάσταση να επαναληφθεί. Ο κύριος ε, Γιαρούς και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη σαφήνεια θα ήθελα να πω ότι το εμπάργο της Ρωσίας, ο αποκλεισμός της Ρωσίας, μας οδηγεί σε μια τριπλή δράση. Πρέπει να έχουμε συνοχή, πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, να δράσουμε όλοι μαζί και να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Η Ρωσία σήμερα θέλει να σπάσει την αλληλεγγύη μας. Δεύτερον, πιστεύω πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πιο στεναρή κατά της Ρωσίας και του αποκλεισμού των ε, οδικών μεταφορών από τη Ρωσία. Τρίτον, πιστεύω θα πρέπει να κοιτάξουμε και πώς μπορούμε να στηρίξουμε οικονομικά όλες αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Χρειάζονται την βοήθειά μας οι μεταφορικές εταιρείες της Ευρώπης μέχρι να σταματήσει ο αποκλεισμός. Πολύ φοβάμαι δεν θα επιβιώσουν μέχρι τότε αυτές οι επιχειρήσεις. Ο κύριος Κουσμούκ έχει το λόγο από την ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στο ότι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Η απόφαση της Ρωσίας είναι η πολιτική απόφαση που ουσιαστικά αποτελεί την απάντηση στις δικές μας κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε τους τομείς αυτούς που σήμερα πλήττονται άμεσα από αυτόν τον αποκλεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα ταμεία που μπορούν να στηρίξουν αυτό το τομέα, ο οποίος πλήττεται από αυτήν την κρίση. Και θεωρώ ότι αυτά τα ταμεία μπορεί να αποζημιώσουν εν μέρη αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Στην Πολωνία το 1 τρίτο του τομέα κινδυνεύει να αφανιστεί κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα πραγματικά να επιστήσω την προσοχή σας στη δραματική κατάσταση που πλήττει τους ε, μεταφορείς από την Πολωνία. Δέχεστε την μπλε κάρτα του τον κύριο Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφε, κάποιοι ήδη αναφέρθηκαν στις ε, αποζημιώσεις. Μπορούμε όμως σήμερα να κάνουμε έναν ε, υπολογισμό για το τι ακριβώς πρέπει να δώσουμε. Ξέρουμε σήμερα ότι μετά τις ε, κυρώσεις υπάρχουν επιπτώσεις και για τους αγρότες. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όλοι σήμερα προσπαθούν να κάνουν ένα απολογισμό. Για το 2014, για την Πολωνία μόνο, οι απώλειες έχουν φτάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλο ποσό και η επιδείνωση της κατάστασης συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν πλήττεται εξίσου και η Τσεχία, αλλά οι βαλτικές χώρες και άλλες πλήττονται. Δεν είναι δηλαδή καθαρά θέμα της χώρες μου. Πρέπει να υπάρξει ανηλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να επιφυλαχθώ ως προς την άποψη ότι οι κυρώσεις δημιουργούν κίνητρα γιατί έχουμε εμπειρία από την Ισπανία του Φρανκό και έχουμε και εμπειρία από την Κούβα. Επομένως οι κυρώσεις σπάνια κατά τη γνώμη μου δημιουργούν κίνητρα. Ωστόσο η Ρωσία πέρσι τον Αύγουστο αποφάσισε να απαγορεύσει εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και αυτό έπληξε ιδιαιτέρως ε, την περιοχή μου που παράγει πεπόνια και βερίκογα καταπληκτικά και τους σταμάτησαν στα ρωσικά σύνορα. Είχαν κάνει χιλιάδες χιλιόμετρων και τελικά τους σταμάτησαν εκεί και τους υποχρέωσαν να γυρίσουν πίσω να αναζητήσουν νέες αγορές ή να χάσουν το φορτίο τους. Μετά από αυτό το συμβάν στα ρωσικά σύνορα ε, επιβλήθηκαν νέες, ε, νέοι όροι στις επιχειρήσεις, ε, κόπηκαν οι εκπτώσεις, αυξήθηκαν οι εγγυήσεις που έπρεπε οι επιχειρηματίες να καλύψουν. Και λέτε εσείς ότι πρέπει οι εμπόροι και οι επιχειρηματίες να βρουν άλλες αγορές. Μακάρι να μπορούσαν σας απαντώ, γιατί και η Γερμανία εφαρμόζει ένα σωρό εμπόδια που δυσκολεύει την ικανότητα των οδηγών να φτάσουν στην αγορά που προορίζονται. Και για τη Γερμανία μπορείτε κάτι να κάνετε και ελπίζω να το πράξετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πυρίνσκι. Παρακαλώ από τους σοσιαλιστές για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να απαντήσετε στο τρίτο ερώτημα που σας απευθύνει ο Πρόεδρος ο κύριος Κράμερ, δηλαδή ποια μέτρα εξετάζει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Και τονίζω η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό που τονίστηκε είναι ότι η Επιτροπή δουλεύει ως ομάδα όχι ο κάθε επίτροπος για τον εαυτό του. Επομένως, όταν λαμβάνεται μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι συνέπειες πρέπει να εξετάζονται από όλους και οι συνέπειες παντού. Εδώ έχουμε τεράστια απώλεια για τους οδικούς μεταφορείς, έχουμε τεράστια διαταραχή της αγοράς και δεν είναι λογική να μας λέτε γυρίστε σπίτια σας και ζητήστε κρατικές ενισχύσεις από τις κυβερνήσεις σας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα προχωρήσουμε στη διαδικασία Catch Ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ, από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Ξέρετε, όποτε υπάρχουν περιορισμοί, πάντοτε κάποιος πλήττεται από αυτό. Απόψε ακούμε πολύ δυσάρεστες ιστορίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν αυτοί οι περιορισμοί και οι κυρώσεις και τον τρόπο με τον οποίο έπληξαν τους μεταφορείς. Ίσως έχει αναφερθεί και νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να συστήσουμε μια επιτροπή για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι θα δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε τι του συμβαίνει. Δεν αρκεί να λέμε ότι θα μπορέσουν τα κράτη να τους βοηθήσουν και τίποτα άλλο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστρέξει. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς τους περιορισμούς, ε, τις απαγορεύσεις μέχρι ότου της άρει η Ρωσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος ε, Πατζήτης από τους σοσιαλιστές. Ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, πράγματι σήμερα ακούσαμε την περιγραφή πολλών προβλημάτων που έχουν πλήξει το τομέα των μεταφορών. Να αναφέρω όμως ότι το θέμα δεν είναι μόνο της οικονομίας των μεταφορών, είναι και πολιτικό ζήτημα, ζήτημα αλληλεγγύης και μου κάνει έκπληξη ότι σήμερα δεν ε, ακούγονται, δεν δίνεται καμία συγκεκριμένη λύση. Ε, συμμερίζομαι βέβαια την κατάσταση σας και καταλαβαίνω πόσο δύσκολε είναι οι συνθήκες που τις οποίες πρέπει να εργαστείτε παρ' όλα αυτά. Πρέπει να ψάξετε να βρείτε κάποιες λύσεις. Καταλαβαίνω τα προβλήματα τη Ιταλία, για παράδειγμα που είχαμε λόγω των μεταναστευτικών ροών κάποια άλλα προβλήματα αλλά και αυτό εδώ είναι πολιτικό ζήτημα. Και το ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχει κάποια αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν απλά θα αφήσουμε τη Ρωσία να συνεχίσει με αυτή την πολιτική του διάρκεια Βασίλευα. Οπότε σας κάνω έκκληση κύριε Επίτροπε να υποστηρίξετε οικονομικά τα κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, η ψυχροπολεμική σύγκρουση ευρωπαϊκής ένωσης ρωσίας έχει προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία του ευρωπαϊκού νότου. στις 9 αυγούστου με ερώτησή μου στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ζήτησα την πλήρη αποζημίωση όχι μόνο των αγροτών της ελλάδας αλλά και των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων. οι έλληνες μεταφορείς έχουν ήδη απολέσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ αφού το 40% των ελληνικών προϊόντων αγροτικών προϊόντων εξάγονται στη ρωσία και μεταφέρονται με φορτηγά. όταν είχε γίνει το εμπάργκο κατά της πρώην ιουγκοσλαβίας το 1992 με τον κανονισμό 525 οι έλληνες μεταφορείς είχαν αποζημιωθεί. τώρα έχω έγγραφο κύριε πρόεδρε εδώ της επιτροπής με ημερομηνία 9 του 2014 που ενημερώνει τους έλληνες μεταφορείς ότι δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι αποζημίωσης από την ευρωπαϊκή ένωση για τη ζημιά που υπέστησαν από το ρωσικό εμπάργκο που ήταν αντίμετρα στα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε η ευρωπαϊκή ένωση. εμπέζει λοιπόν η ευρωπαϊκή ένωση και η επιτροπή τους έλληνες μεταφορείς καλώντας τους μόνοι τους να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους το οποίο αντιμετωπίζουν. κρίμα κύριοι της επιτροπής. Ευχαριστώ. Ε, E, Κύριε Βόλτς, έχω μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να νοστοποιώσουν στη Ρωσία την κατάσταση. Νομίζω πραγματικά ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει εδώ να υιοθετήσουν μια κοινή στάση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτές που και στις μεταφορές και στον αγροτικό τομέα έχουν πληγεί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αποκλειστικά για τον ένα ή τον άλλο τομέα. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση συνολική. Γιατί οι κυρώσεις αυτές μπορεί να συνεχιστούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα πρέπει οπωσδήποτε η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο να αναφερθούν συνολικά στο θέμα αυτό. Ο κύριος Φεραίρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι οδικοί μεταφορείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πληγεί από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία έχει να κάνει και με τις παράπλευρες ζημιές λόγω της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, θέσεις απαράδεκτης ε, που οδηγεί σε εμβάθυνση της ρήξης και που δεν έχει λάβει υπόψη τις οικονομικές, ε, πολιτικές, γεωστρατηγικές επιπτώσεις. Λόγω ανομολόγητων συμφερόντων έχει αποσταθεροποιηθεί η Ουκρανία, έχουν προωθηθεί νεοναζιστικές δυνάμεις ε, και τώρα λέμε ότι υπερασπιζόμαστε τα ε, συμφέροντά μας. Σε αυτό το πλαίσιο διάφορες επιχειρήσεις ε, μεταφορών υδατοκαλλιέργειας αλίας υποφέρουν από τις παράπλευρες ζημίες σε αυτή τη στρατηγική υπεράσπιση άλλων συμφερόντων. Δεν μπορείτε να ανέβετε τα σχέδια σας έτσι. Έχετε άμεση ευθύνη για αυτές τις ζημίες και δεν μπορείτε απλά να συζητάτε πιθανές ε, αποζημιώσεις που θα καταβάλουν ενδεχομένως τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον πρόεδρο τον κύριο Κράμερ, ε, ναι, πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών. Παρακαλώ κύριε Κράμερ. Κοιτάξτε, η Ρωσία το 1994 παραβίασε της τη Βουδαπέστης. Και φυσικά, ενώ διασφάλισε την ε, εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, είδαμε πώς αντέδρασε η Ρωσία. Η Ρωσία παραβίασε αυτήν την συνθήκη και οι, συν, οι κυρώσεις οι δικές μας ήταν συνέπεια και αντίδραση σε αυτήν την παραβίαση. Ναι ή όχι. Ήταν έγκλημα αυτό που έκανε η Ρωσία. Ναι ή όχι. Αγαπητέ κύριε Κράμερ, να απαντήσω στην ερώτησή σας με μια άλλη ερώτηση. Κοιτάξτε ένα τμήμα της ιστορίας. Δεν κοιτάτε ολόκληρη την ιστορία. Κύριε Κράμερ, ξεχάσατε τις δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της κυρίας Νιούλαντ, Υπουργού Εξωτερικών, όσον αφορά τις δυνάμεις τις ναζιστικές, τις φασιστικές που έχουν αναλάβει την εξουσία στην Ουκρανία. Και βέβαια το πραξικόπημα που έγινε εκεί υποστηρίχθηκε από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, παρόλο που η ρωσική απαγόρευση προκάλεσε τεράστιο πλήγμα στις οδικές μεταφορές. Ο κλάδος αυτός δεν έτυχε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο μάλιστα. Η Γαλλία και το Βέλγιο επέβαλαν νέα μέτρα ως προς το, την περίοδο ανάπαυσης των οδηγών. Η, Γερμανία θεσμοθέτησε το βασικό μισθό. Όλα αυτά χρησιμεύουν στις τοπικές επιχειρήσεις και πλήττουν και μάλιστα πολύ τους μεταφορής των χωρών της Βαλτικής. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να αποζημιώσετε τον κλάδο των μεταφορών στις χώρες της Βαλτικής και καλό το, τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία να παραιτηθούν από αυτά τα μέτρα που αποτελούν διάκριση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Χέτμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα του πώς το ρωσικό επάρκο έπληξε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το κόστος ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, το γνωρίζουμε όλοι, και ο αντίκτυπος γίνεται αισθητός στον κλάδο των μεταφορών, αλλά όχι μόνο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει αλληλεγγύη και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις ε, μεταφορικές επιχειρήσεις της Ευρώπης. Ίσως θα πρέπει να δεχθούμε τις αρχές της ε, ενίσχυσης θα πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε όλα αυτά, θα μας βοηθήσουν και να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το καθεστώς. Ευχαριστώ κύριο Βοητσιχόφσκι από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναμφισβήτητα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποζημιώσει, να καλύψει το κόστος που υπέστησαν όλοι αυτοί που πλήττονται, που υποφέρουν λόγω αυτών των απαραίτητων κυρώσεων. Και εμένα με σόκαρε αυτό που είπε ο κύριος Φερέιρα, ξέρετε. Μιλάτε για νέο φασίστες στην Ουκρανία και λέτε ότι οι δράσεις μας είναι το αποτέλεσμα των δικών τους δράσεων. Νομίζω ότι δεν ξέρετε τι γίνεται εκεί πέρα. Η Πορτογαλία είναι πάρα πολύ μακριά και ενδεχομένως γι' αυτό δεν έχετε παρακολουθήσει σωστά τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ είναι μια τεράστια απειλή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ε, αντιμετωπίζουμε την προπαγάνδα του Κρεμλίνου και λυπούμε πολύ που σας άκουσα να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να ζητήσω τώρα από την κυρία Επιτρόπο να απαντήσει στις πολυάριθμες παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών που ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια αντίδραση, κάποια βοήθεια. και όχι να ρίχνει τις ευθύνες ε, ε αντιμετώπιση του προβλήματος στα κράτη-μέλη. Και ουσιαστικά εδώ αναρωτιόμαστε κατά πόσο οι μεταφορικέ εταιρείε θα μπορούσαν να λάβουν κάποια ε, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, κύριε Επιτρόπε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Κατέγραψα όλες τις ανησυχίες και θα φροντίσω να λυθούν υπόψη από την Κομισιόν ε, στις σημερινές της εργασίας. Επίσης υπόσχομαι ότι θα εξετάσουμε τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που κάνατε έγκαιρα έχω επίγνωση του γεγονότος ότι όλα σε αυτές τις προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με οριζόντιο τρόπο. Τα πράγματα είναι σοβαρά και επικίνδυνα. Να επαναλάβω ότι η Κομισιόν συμμερίζεται τις ανησυχίες ε, όσον αφορά τις οικονομικές ζημίες ορισμένων επιχειρήσεων λόγω του ρωσικού εμπαργού. Η Κομισιόν εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση αναμένουμε ανάλυση στο άμεσο μέλλον. Την παρουσία στιγμή δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία για σημαντικές, ε, σημαντικά προβλήματα στην αγορά πέραν κάποιων ε, μεμονωμένων περιπτώσεων όσον αφορά το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης που αναφέρθηκε. Ε, αυτό έχει σκοπό να υποστηρίζει απολυμμένους εργαζομένους όπως έχει σήμερα δεν έχει σχεδιαστεί για να παράσχει αποζημιώσεις ε, λόγω ζημιών ε, σε περιπτώσεις όπως αυτή που συζητάμε σήμερα συγκεκριμένα το ρωσικό εμπάργο. Το το που έχω να πω, τα ανακουφιστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο είναι δυνατά, αλλά πρέπει να ακολουθούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να αξιολογήσει οποιαδήποτε προγράμματα προβλεφθούν σε εθνικό επίπεδο. Ξέρω ότι αυτή τη λύση δεν είναι τέλεια, αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικό της προπολογισμό για να βοηθήσει ε, την ε, πολιτική μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο περιορισμένα μέσα για δράσει ε, στο πλαίσιο τη εξωτερική πολιτική. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν στενά με τα κράτη-μέλη για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τι σοβαρότερε ε, συνέπειε δράσεων από τρίτε χώρε. μια ταχεία και μακροπροθεσμή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ευρώπη και Ρωσίας θα ήταν φυσικά επιθυμητή αλλά στην παρουσία φάση το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι ότι η πολιτική κατάσταση θα βοηθήσει τις προσπαθίες μας συντομότερο δυνατόν. Ναι, πρέπει όντως να κάνουμε κάτι. Θα συνεργαστώ λοιπόν με εσάς και τα κράτη-μέλη ώστε να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε ενδεχομένω να καταλήξουμε σε νέε πιθανέ λύσει με τον ΠΟΕ. Αυτό θα είναι το πρώτο σημαντικό μα βήμα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση ενώ εξελισσόταν προσπάθησα να πάρω το λόγο γιατί η Αυστρία πραγματικά επηρεάζεται από όλη αυτή την κατάσταση. Δώσατε το λόγο σε πολλούς συναδέλφους, αλλά όχι με ισορροπημένο τρόπο. Πολλές κυρίες και κύριοι από το δικό σας κράτος πήραν το λόγο και εγώ προσπάθησα πολλές φορές και δεν μου τον δώσατε, ενώ και η δική μου χώρα πλήττεται. το όνομά σας ήταν στον κατάλογο. Ζητώ συγγνώμη, δεν το είδα. Εγώ φταίω. Πραγματικά σας ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ την ε, Επίτροπο.